Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης με την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά την ημερησία διάταξη. Όχι, εγκρίνεται επομένω. Στο φακελό σας έχετε λάβει τις συστάσεις και τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των συντονιστών το ης Σεπτεμβρίου. Αν ε, έχετε παρατηρήσεις για το αποτέλεσμα αυτής της συνεδρίασης, να το πείτε στη γραμματεία πριν από το τέλος ε, της σημερινής συνεδρίασης. Διαφορετικά, θεωρείτε ότι εγκρίνονται. Έχω μία ανακοίνωση από πλευράς μου. Θα ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας τις εντυπώσεις και τα αποτελέσματα του τελευταίου μου ταξιδιού στην Καμπούλ, στο Αφγανιστόν. Γύρισα στο βράδυ. Ξέρετε ότι εκεί ε, η δουλειά μου έχει να κάνει με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεν προχωρούν καλά οι εργασίες, μπορούμε να το πούμε, σε ό,τι αφορά το φάκελο της Καμπούλ σε σχέση με τις τράπεζες. Ε, βρήκαμε πάνω από 600 πάνω από 6 καταδικασμένους και 29 άλλα άτομα για τα οποία πρέπει να αρχίσουν έρευνες, όμως δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι έρευνες αυτές. Ο Γενικός εισαγγελέα. δεν είναι πολύ ενεργητικός. Επίσης υπάρχει ένας ακόμη μεγάλος φάκελος ε, για διαφθορά, υποψίες για διαφθορά 42 εκατομμυρίων δολαρίων που έπρεπε να δοθούν στο στρατιωτικό νοσοκομείο και δεν βρίσκουμε ίχνος από αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, η ε, ιδέα ότι κάποιος έκλειψε τα φάρμακα που προορίζονταν για τους στρατιώτες μιας χώρας μου δείχνει πόσο παρούσα είναι η διαφθορά και πόσο μεγάλη είναι η ατιμορρησία. Ε, κατά τα λοιπά προετοιμάζονται οι εκλογές για τον Απρίλιο του 2014 θα υπάρχουν προεδρικές εκλογές ε, στο Αφγανιστάν και οι εγγραφές των υποψηφίων ε, θα ολοκληρωθούν στο τέλος της εβδομάδας. Μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί τέσσερις υποψήφοι και το σύστημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Χρειάζονται 5.000 υπογραφές ε, και με την ταυτότητα, τον αριθμό ταυτότητας για να μπορεί κάποιος ε, να θέσει υποψηφιότητα και υπάρχει μια ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή η οποία εργάζεται πολύ σκληρά όμως ε, επειδή υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας σε ολόκληρη χώρα αυτό κάνει πολύ δύσκολο να καταρτιστούν οι εκλογικοί κατάλογοι. Όμως ε, θεωρούνται αυτές οι εκλογές πάρα πολύ σημαντικές ε, από όλους ε, όσους συνάντησα. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί ακόμη. Η απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων στα πλαίσια αυτής της αποστολής στο τέλη του 2014 υπάρχουν τρέχουσες διαπραγματεύσεις για να δούμε υπό ποιες συνθήκες τα αμερικανικά στρατεύματα ή ένα τμήμα τους μπορούν να μείνουν μετά το 2014 και περιμένουμε την ε, ολοκλήρωση μιας συμφωνίας, τη σύναψη μιας συμφωνίας. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από το Αφγανιστάν, ολόφρεσκα. Εκεί δεν ε, έχει βελτιωθεί, δεν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες ασφαλείας στην πραγματικότητα όπως γνωρίζετε. Παρακαλώ από την Κομισιόν. Όχι, ο κύριος Μαρτίνες. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα ένα λεπτό να αναφερθώ στα πρακτικά της συνεδρίασής μας ε, στο θέμα αυτό, στο σημείο αυτό. Μόλις ε, επιστρέψαμε από τη Νέα Υόρκη, εγώ ήμουν μέρος αυτής της αποστολή είναι προφανές ότι θα καταρτιστεί μια έκθεση για αυτή την αποστολή, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, αλλά πιστεύω ότι είναι ήδη καλό, όπως κάνατε κι εσείς, να σημειώσουμε ότι στη συνεδρίασή μας κάτι θα υποθεί σχετικά. Καταρχήν, θέλω να υπογραμμίσω την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την φιλικότητα με την οποία ο κύριος Κασμάρεκ προείδρευσε της αντιπροσωπείας. Το πρόγραμμα ήταν ενδιαφέρον συναντήσαμε και τον πρόεδρο της Παγκοσμίας Τράπεζας αλλά και υψηλά ηθήνοντες του προγράμματος του ΙΕ για το περιβάλλον και, για το περιβάλλον και συζητήσαμε την υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας. Ήταν ενδιαφέρον λοιπόν το πρόγραμμα. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι η διάσκεψη για την ανάπτυξη και για την υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας ήταν πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι προσδοκούσαμε. Και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι οι σχέσεις ε, που δημιουργήθηκαν δείχνουν ότι έχουμε προχωρήσει περισσότερο προς την υλοποίηση των στόχων από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί, ναι, μεν ε, παραπονιόμαστε για όσα παραμένουν να γίνουν, αλλά αυτό μπορεί να υποτιμήσει, να οδηγήσει σε υποτίμηση των όσων έχουν ήδη επιτευχθεί. Η διάσκεψη ήταν ενδιαφέρουσα και ακούσαμε κάποιες φωνές πάρα πολύ σημαντικές. Ο δεύτερος ομιλητής ήταν ο κύριος Μπαρόσο άλλωστε, ο οποίος μίλησε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξ ονόματος όλων μας δηλαδή. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τα πούμε αυτά για να τα έχουμε υπόψη και δεν θα παραπανεθώ παρά για ένα πράγμα ότι με την ευκαιρία αυτής της διάσκεψης για την υλοποίηση των στόχων της χιλιτίας ο, υπήρχαν μόνο άνδρες στο Προεδρείο και όσοι πήραν το λόγο ήταν μόνο άνδρες. Ενώ Όλοι αναγνωρίζουν τη μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει σε θέματα που αφορούν τις γυναίκες. Εγώ ομολογώ ότι αν η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αποτελούταν από εννέα άνδρες και είχαμε και κάποια γυναίκα στην μέσα προσωπία, θα, νιώ, θα νιώθα καλύτερα όπως είπα, γιατί και εγώ ένιωθα λίγο άσχημα να σκήσω κριτική για την έλλειψη των ε, γυναικών. Όμως ε, ξέρετε πως ε, στελεχώνονται οι αντιπροσωπείε μας, δεν ευθύνεται κανείς, όμως θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε αυτά. Γιατί τελικά αυτό οδηγεί σε αποδυνάμωση των όσων διεκδικούμε σε τόσο σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μαρτίνες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρτίνες που αναφερθήκατε σε αυτό το σημαντικό γεγονός και τονίσατε πόσο σημαντικό είναι να δουλεύουμε πάντοτε για τους στόχους της χιλιετίας Κατά τη διάρκεια τη σημερινή μα συνεδρίαση θα μιλήσουμε για τον Μπαγκλαντέ. Να καλωσορίσω επί τη ευκαιρία και του προσκεκλημένου μα που θα μιλήσουν για τη σημασία των στόχων αυτών για εκείνου. Όπω επίση θα μιλήσουμε και για το πράσινο ακροτήρι και θα δείτε ε, πώ ε, επέτυχαν του στόχου τη χιλιετίας δεν υπάρχουν ερωτήσεις, οπότε να περάσουμε στο πρώτο ουσιαστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, την κλιματική αλλαγή ε, από την οπτική γωνία του Παγκλαντές. Η ανταλλαγή απόψεων ε, θα αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή και η συζήτηση δεν θα μπορούσε να ε, συμβαίνει σε καλύτερο ε, σημείο χρονικά, γιατί την περασμένη εβδομάδα η κυβερνητική ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κλιματική αλλαγή ε, δημοσίευσε την έκθεσή της. Σήμερα δημοσιεύει την έκθεση αξιολόγησή της, αξιολόγησής της ε, για τα πιο σημαντικά συμπεράσματα για την κλιματική αλλαγή από το 2007. Γιατί κάθε έξι χρόνια δημοσιεύεται η έκθεση αυτή. Βάσει επιστημονικών ε, στοιχείων όσο το δυνατόν πληρέστερων, η έκθεση αξιολόγησης παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το κλίμα θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ κρίσιμος ο ρόλος αυτός. Ο, η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και στη δική μας Επιτροπή. Σήμερα το απόγευμα θα ε, ψηφίσουμε... Ε, μία... θα ψηφίσουμε και ένα σχετικό θέμα στην ε, ημερήσια διάταξή μας, τη διάσκεψη των ΗΕ για την αλλαγή του κλίματος στη Βαρσοβία. Θα θέλαμε λοιπόν να ε, ακούσουμε τις απόψεις ε, του ε, Μπαγκλαντές, δεδομένου ότι πλήττεται ιδιαίτερα από την επίδραση της αλλαγής του κλίματος και θα επιδεινωθεί η κατάσταση πλήττοντας τα δέλτα των ωκεανών, παράκτιες περιοχές, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Μπαγκλαντές. Θα μας πείτε πόσα άτομα ε, ζουν ε, σε εσά ε, στον στο δέλτα του ποταμού. νομίζω ότι είναι 10 εκατομμύρια περίπου, αλλά εσείς θα μας το πείτε. Θα ακούσουμε λοιπόν πολύ προσεκτικά τους ε, αντιπροσώπους του Μπαγκλαντές να μας εξηγήσουν πώς ε, ε, βλέπουν την αλλαγή του κλίματος, πόσο είναι ευάλωτη η χώρα, η τους και τι ελπίζουν, από ποιες είναι οι προσδοκίες τους από τη Βαρσοβία. Επιτρέψτε μου εκ μέρους της ομάδα, της Επιτροπής μας να καλωσορίσω τον ε, ε, κύριο Αζαντούζαμαν, ε, ο οποίος είναι, συμμετέχει στους, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις εδώ και 10 χρόνια, τον Αξάντου Χάμεντ που είναι ερευνητή για το κλίμα και συμμετέχει στις διεθνείς διαπραγματεύσεις από την αρχή των διαπραγματεύσεων αυτών, τον κύριο Καμρούλ Τσαουντουρί, μέλος της Επιτροπής Προσαρμογής που συστήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές, Γενικό Γραμματέα του ε, World Water Forum of Journalists. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Νομίζω δύο παρουσιάσεις θα γίνουν και προτείνω στη συνέχεια οι ευρωβουλευτές να έχουν τη δυνατότητα να σας θέσουν ερωτήματα και να κάνουν σχόλια σας ε, αφήνω να αποφασίσετε ποιος θα κάνει την πρώτη και ποιος τη δεύτερη παρουσίαση. Περίπου 8 λεπτά έκαστη. Έχετε το λόγο λοιπόν. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω την εισαγωγή στο θέμα και στην αδελφή μου θα ακολουθήσουν αργότερα. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, ας ε, ξεκινήσω απευθείας με την ουσία του θέματος, χωρίς να μακρηγορήσω. Υπάρχουν δύο θέματα από δύο, δύο διαφορετικές σκοπιές. Τι μας λένε οι επιστήμονες για το κλίμα και τι προσδοκίες έχουν οι άνθρωποι. Κάποιος γνωστός ποιητής μας είπε ότι τα δέντρα, κάποιος επιστήμον ερευνητής μάλλον, μας, είπε, μας λέει ότι ένα συγκεκριμένο είδος δέντρο ανθίζει ε, την άνοιξη, αλλά τώρα ανθίζει ε, συνέχεια και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Όλα αυτά οφείλονται κατά κάποιο τρόπο της, ε, στην αλλαγή του κλίματος. Καινούργια φαινόμενα, καινούργιες... Ε, αποδείξεις και ενδείξεις από την επιστήμη, όπως έχουν προκύψει συμπεράσματα από την ομάδα εργασίας 1 του IPCC. Όλα αυτά τα συμπεράσματα και οι ενδείξεις μας δείχνουν το εξής. Πρώτον, ότι υπάρχουν εποχές πρόσφατες όπου η άνοδος της θερμοκρασίας στη γη έχει, έχει μειώσει το ρυθμό της. Αυξάνεται με πιο αργό ρυθμό. Ε, αυτό ισχύει και για τους βαθείς ωκεανούς. Η θερμοκρασία των ωκεανών αυξάνεται και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και ανησυχητικό. Ποιες ε, είναι τώρα οι επιπτώσεις από, αυτές, από όλα αυτά τα φαινόμενα και τι ακριβώς επιπτώσεις υπάρχουν στο Μπαγκλαντές η, Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μπαγκλαντές πρόσφατα άρχισαν να συνεργάζονται και υπάρχουν νέες πτυχές, νέοι τομείς στους οποίους η συνεργασία είναι απαραίτητη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μπαγκλαντές θα πρέπει να στοχεύσουν στη συνεργασία και σε αυτούς τους άλλους τομείς την άδεια της Προέδρου του Προεδρείου ε, θα ήθελα να ε, διανύμω ένα φυλάδιο το οποίο ε, αναφέρεται συγκεκριμένα στην κλιματική αλλαγή και να δώσω το λόγο, μου, το λόγο στο συναδελφό μου. Thank you. Να μιλήσει περισσότερο για αυτό το θέμα. Κυρία Πρόεδρε, είμαι ε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, αξιότιμα μέλη κυρίες και κύριοι, το Μπάγκλα είναι μία από τις λιγότερο χώρες και έχει κάνει σημαντική πρόοδο σχετικά με την άμβλυνση της φτώχειας ε, και έχει προσπαθήσει έντονα να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, να μειώσει την παιδική θνησιμότητα ε, και μητρική θνησιμότητα ε, τα τελευταία χρόνια και επίσης να θέσει τα θεμέλια μιας, μιας κοινωνίας που να βασίζεται στην ισότητα και στην δικαιοσύνη και επίσης να εντάξει όλα τα κορίτσια τουλάχιστον στο, σε δημοτικά σχολεία. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, το Μπαγκλαντές πιστεύουμε ότι θα περάσει από τις λιγότερο αντιγμένες χώρες σε, ανε... σε ε, αναπτυσσόμενες χώρες προς τα μέσα του, του 2021 ε, που θα συμπέσει κατά κάποιο τρόπο με την πεντηκοστή επέτειο της ανεξαρτησίας του. Τώρα όμως με όλες τις προσπάθειες αυτές που κάνουμε αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή ε, την ε, ε, μείωση των πηγών ίδρευσης και του, του, του νερού, του, του νερού ως πηγής ζωής, την, τα μεγάλα προβλήματα στη γεωργία, στην ασφάλεια των τροφίμων, σε μια χώρα που μην ξεχνάτε αριθμεί 160 εκατομμύρια κατοίκους. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, η οποία τόσα πολλά έχει επενδύσει στην αναπτυξιακή προσπάθεια αυτής της χώρας ε, θέλει να παραμείνει η κατάσταση ως έχει, δηλαδή με όλες αυτές τις ενδικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι όλη αυτή η πρόοδος την οποία έχουμε επιτύχει θα διαλυθεί, θα καταρρεύσει, αν συνεχίσουμε έτσι. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να εξηγήσω σε φάσεις πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τη ζωή μας. Ήδη η γεωργία απειλείται, επειδή αυξάνονται συνέχεια και γίνονται και πολύ πιο σοβαρές οι πλημμύρες. Ε, αυξάνονται η βροχή, η συχνότητα των βροχών και η δύναμη των βροχών και επίσης ε, οξύνονται οι ξηρασίες η θερμοκρασία αυξάνεται, η γη ξεραίνεται ε, και αυξάνεται και το περιεχόμενο σε, σε αλάτι της ε, γης. wave interactions due to ε, και στις παράκτιες περιοχές. Οι παράκτιες περιοχές απειλούνται συνέχεια από κυκλώνες, από τυφώνες και από τσουνάμι, ε, δεδομένου ότι υπάρχει μια σαφής διασύνση μεταξύ αύξησης της θερμοκρασίας και ε, πλημμυρίδων και επηρεάζουν εκατομμύρια ζωές που ζουν από την αλία στις παράκτιες περιοχές. Η ασφάλεια των τροφίμων μαζί με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, όπως η, αύξηση της αλμυρότητας του νερού ε, και η αύξηση παθοόνων ε, μικροβίων και μολυσματικών ασθενειών, θα επηρεάσουν την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων, εκατομμυρίων κατοίκων, ιδίως αστικές περιοχές, επειδή εκεί υπάρχει τεράστια πυκνότητα πληθυσμού. Γι' αυτό προβλέπεται ότι ο μισός πληθυσμός μέχρι το 2030 θα κατοικεί σε αστικές περιοχές. Δηλαδή, ε, οι μισοί κάτοικοι του Μπαγκλαντές θα μένουν σε αστικές περιοχές στα μέσα του, ε, γύρω στο 2030 που ε, ως αποτέλεσμα δηλαδή της μετατόπισης του πληθυσμού και της εξόδου από την Ήπεθρο προς τις πόλεις. Όσον αφορά τώρα τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις, δεν μπορούμε να συζητήσουμε την κλιματική αλλαγή χωρίς να λάβουμε υπόψη και τις οικονομικές πτυχές. Σε μερικές ε, περιπτώσεις γίνεται δύσκολο να σχεδιάσουμε αναπτυξιακά έργα χωρίς, επειδή ακριβώς υφίσαν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σε άλλες περιπτώσεις η χρηματοδότηση έργων ε, απαιτεί μία προσαρμογή σε εντελώς νέους τομείς και νέες δραστηριότητες λόγω της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων. Παραδείγματο χάρη, η ανάπτυξη, ε, η ανάπτυξη ενός ε, καινούριου προηγμένου τεχνολογικά σπόρου ριζιού στην οποία επιτύχαμε, επιτρέπει μια συχνότερη εσοδεία, αλλά δυστυχώς η καινούργια αυτή εσοδεία και όλη αυτή η προσπάθεια ξαναμίζεται λόγω της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Οι επιστήμονες του Μπαγκλαντές έχουν ήδη επιτύχει να αναπτύξουν κυριότερες ε, ε ποικιλίε ε, ε, σπόρων, ποικιλίε ριζιού κυρίω, οι οποίε με, περισσότερε εσοδίε κατά τη διάρκεια του χρόνου και λιγότερη αρμυρότητα. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα έργα για να δώσουμε στους αγρότες και στους πραγούς τη δυνατότητα επιλογών και ελευθερίας. Όπως συμφωνείται η ελευθερία επιλογών συνάδει με την ανάπτυξη. Ήδη διανύουμε το έκτο πενταετές ε, πρόγραμμα ε, προσπαθώντας να ενσωματώσουμε τις κλιματικές αλλαγές στα αναπτυξιακά έργα. Ε, αυτή η αλλαγή πολλές φορές απαιτεί νέες πιστώσεις, νέες χρηματοδοτήσεις πέραν των τακτικών και σε ορισμένες ε, περιπτώσεις τα προγράμματα αυτά δεν θα είχαν ξεκινήσει, δεν θα υπήρχε δηλαδή το επιπλέον κόστος εάν δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή. Τώρα αν αυτό το λέτε στις πληρωματικές δαπάνες ή όχι δεν ξέρω, πάντως η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη στην πραγματικότητα. Υπάρχει η ανάγκη χρηματοδότησης, όπως είπα, νέων μορφών δραστηριοτήτων. Μία από τις μορφές αυτές είναι οι, οι, οι μελέτες κόστους-οφέλους και οι μελέτες ε, ζημιών λόγω των επιπτώσεων του κλίματος. Ε, οι άνθρωποι όμως αναγνωρίζουν το πρόβλημα και δεν ε, κάθονται μυρολατρικά να υφίστανται τις επιπτώσεις. Οι αγρότες παραδείγματο χάρη ε, σε όλο τον κόσμο και στο Μπαγκλαντές προσπαθούν να βρουν τρόπους προσαρμογής. Ποιος όμως θα τους αποζημιώσει για τα επιπλέον τις επιπλέον δαπάνες τις οποίες ήδη έχουν πληρώσει, καταβάλει. Η αποζημίωση για τις ζημίες και τις αρνητικές επιπτώσεις πρέπει να καλυφθούν από τα κεφάλαια ε, ζημιών και απολειών. Αυτό είναι ένας νέος τρόπος ε, κλιματικής χρηματοδότησης, αν θέλετε, η οποία ξεπερνάει την αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Το άλλο πρόβλημα είναι βεβαίως πώς μπορούμε να μειώσουμε το, τους κινδύνους, το, το ρίσκο και να εφαρμόσουμε μηχανισμούς μείωσης του κινδύνου. Ποιος θα πληρώσει όμως όλα αυτές τις ε, δαπάνες. Οι αγρότες στο Μπαγκλαντές έχουν ελάχιστες χρηματοδοτικές ε, δυνατότητες. Το, η κυβέρνηση θα το σηκώσει αυτό το τεράστιο κόστος. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα νέο είδος χρηματοδότησης το οποίο ε, χρειάζεται, το οποίο δεν έχει ακόμα ε, βρεθεί, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί και να αποκαλείται climate financing μαζί, δηλαδή με το development, με την χρηματοδότηση ε, για ανάπτυξη, αναπτυξιακή χρηματοδότηση, να υπάρχει και κλιματική χρηματοδότηση θα κάνουμε μια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει την γρήγορη ανάπτυξη δυναμικού στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στις λιγότερο ε, ανεπτυγμένες χώρες από τα αναπτυσσόμενες όπως το Μπαγκλαντές, διαθέτοντας πιστώσεις ταχύτατα. Αναγνωρίζουμε τη καλή συνεργασία και την ε, στήριξη που έχει προσφέρει στο Μπαγκλαντές και πιστεύουμε ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μειώσουμε τους κινδύνους, το ρίσκο και να βελτιώσουμε τον ε, το δυναμικό ε, αναπτυξιακών υποδομών και πλαισίων για να αντιμετωπίσουμε τη κλιματική αλλαγή στο Μπλαγκλαντές. Είναι σαφές ότι υπάρχει, είναι, είναι επίγουσα η φύση της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Ε, πρέπει να δράσουμε με... Είναι ένα επίγον θέμα και Δυστυχώς ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ τον Μπαγκλαντές και άλλες χώρες να προσαρμοστούν στις νέες αυτές συνθήκες. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί αυτή της προσπάθειας, να διαδώσει το μήνυμα και να ε, ε, ακολουθήσει τα συμπεράσματα του IPCC ως παράδειγμα και να πρωτοστατήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια διεθνώς και δι για τον Μπαγκλαντές. Έχουμε επίσης μπορέσει να υλοποιήσουμε τα, τους στόχους άμβλησης των ε, αρνητικών επιπτώσεων. Έχουμε ένα, είχαμε ένα εφταετές πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε νωρίτερα από τη λήξη του. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα φιλόδοξο νέο πρόγραμμα άμβλησης του ρίσκου ε, και των κινδύνων το 2014. Επίσης χρειάζεται περαιτέρω παγίωση των συμπερασμάτων του, του Durban και να καθίσουμε μαζί με το IPCC για να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να καταλήξουμε σε, νομικά ε, σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ε, στο Παρίσι. Η COP19 θα γίνει σε, 19, σε λίγες μέρες στην Βαρσοβία. Βαρσοβία και ε, βεβαίως γίνεται εντός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα θέλαμε, κυρία Πρόεδρε, να ενσαρρύνουμε την, και να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να, να ηγηθεί αυτής της μεγάλης προσπάθεια για να μπορέσουμε και εμεί να επιτύχουμε του στόχους μας και να δικαιωθούμε για όλες αυτές τις προσπάθειες που κάναμε τις τελευταίες δεκαετίες. Ιδίω μετά από την συνεργασία την οποία παγιώσαμε στο Durban με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να με ακούσετε. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε με τον ε, κύριο Τσαουτχάρη. Έχετε και άλλο χρόνο στη διάθεσή σας, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Okay. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα όσα επεσήμαναν οι δύο αξιότιμοι συνάδελφοι καλύπτουν γλαφυρά όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να τονίσουμε. Όλοι ξέρετε ότι στον Τέρμπαν είχαμε δημιουργήσει μια ουσιαστική συμμαχία η λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν όλες τους τις δυνάμεις του Ντάρμπαν για να προωθήσουν μία δεσμευτικά νομική συμφωνία που θα συνεχθεί από όλα τα μέρη, από όλες τις χώρες, από όλες τις υπήρους. Γιατί η άμβληση, ο μετριασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και επίσης αυτό υπόθηκε και από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, την Παρασκευή στη Σοχόλμη. Έτσι λοιπόν, ακούστηκε με σαφήνεια ότι θα πρέπει να αναλάβουμε άμεση δράση για να αναχαιτήσουμε τις παγκόσμιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχει ένα μέτωπο μετριασμού λοιπόν των εκπομπών και στη Βαρσοβία πρέπει να συμφωνήσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε όσο δυνατόν καλύτερα αυτό το θέμα της μείωσης των εκπομπών δηλαδή με έναν τρόπο όπου θα συμμετέχουν όλα τα μέρη. Θα πρέπει επίσης στη Νέα Συμφωνία που ελπίζουμε να υπογραφεί στο Παρίσι το 2015 να συμπεριλάβουμε το θέμα της προσαρμογής, γιατί η προσαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως για χώρες όπως το Μπαγκλαντές, που είναι οι πλέον ευάλωτες. Έτσι λοιπόν, ε, όσο περισσότερο κάνουμε τώρα, τόσο λιγότερο θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε. Αν μειώσουμε τις εκπομπές μας, ε, τότε ενώσουμε λιγότερο τι εκπομπέ μα, με συγχωρείτε, θα πρέπει να προσαρμοστούμε περισσότερο. Όμω υπάρχουν και κάποια όρια, Πρόεδρε. Γι' αυτό πρέπει να επιτεχύνουμε τι προσπάθειε του μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και αν ε, οι φιλοδοξίε μα είναι μεγαλύτερε, τότε δεν θα πρέπει να περάσουμε στην προσαρμογή. Αλλά και ιστορικέ εκπομπέ επίση προκαλούν κάποιες απαιτήσει προσαρμογής. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε αυτές τις ανάγκες προσαρμογής και να βρούμε και την κατάλληλη χρηματοδότηση για την προσαρμογή και πρέπει να έχουμε και οικοδόμηση δυνατοτήτων και μεταφορά τεχνολογίας. Όλο αυτό πρέπει να καλύπτεται από το Global New Deal του 2015 και ελπίζω ότι όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα εντάξουμε σε μια νέα δεσμευτική συμφωνία που θα ισχύει σε διεθνές επίπεδο και ελπίζω να έχει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει ιστορικά ζωτικό ρόλο, όχι μόνο το 1991 και 92 με την με την εκπόνηση της ίδιας της συμφωνίας, εξακολουθώ να θυμάμαι ότι το Μάιο του 1992 η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και τότε χώρες όπως το Μπαγκλατές είχαν συμμετέχει σε αυτή τη συμμαχία. Και από εκεί και πέρα επίσης ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε ηγετική θέση. Και επίσης και στο Κιώτο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πιο ευάλωτες χώρες είχαν ηγετικό ρόλο. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να πράξουμε και στη Βαρσοβία έτσι ώστε να πετύχουμε αυτή την παγκοσμία συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Θα δώσω και εγώ μια ερώτηση. Θα ήθελα να μας πείτε, να κατανοήσουμε καλύτερα πόσο ευάλωτο είναι το Μπαγκλαντέ στην κλιματική αλλαγή, όχι δηλαδή με αφηρημένου όρου, αλλά να μα πείτε συγκεκριμένα τι συμβαίνει, τι παθαίνουν οι άνθρωποι όταν, ε, ε παραδείγματο χάρη, έχουμε τέτοιες πλημμύρες ε, και πόσοι θίγονται στο Δέλτα και πώς τα καταφέρνουν σήμερα, πόσοι πλήττονται εκεί στο Δέλτα. Μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που ζουν στο Δέλτα. και ποιες είναι οι συνέπειες της αύξησης του επίπεδου της θάλασσας. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η ζωή και η περιουσία ή τα υπάρχοντα των ανθρώπων που ζουν στις παράκτιες περιοχές βρίσκονται σε μια πάρα πολύ ευάλωτη κατάσταση για την οποία δεν φταίνε καθόλου. Υποφέρουν όμως τώρα υπό το βάρος αυτών των φαινομένων. Τουλάχιστον 22 εκατομμύρια άνθρωποι, το λιγότερο 22 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν στις παράκτιες περιοχές πόσιμο νερό, διότι ακόμα και τα υπόγεια ύδατα και ο υπόγειος ε, ορίζοντας των υδάτων ε, είναι μολυσμένος. Τι είναι? Γίνεται υφάλμυρος. Είναι υφάλμυρος. Και παρόλα αυτά χρησιμοποιούν, πρέπει να περπατήσουν πολλά ε, μίλια για να βρουν νερό το οποίο είναι λιγότερο υφάλμηρο για να χρησιμοποιήσουν στις καθημερινές τους ε, δουλειές και να γεμίσουν ένα δοχείο. Αυτές είναι οι δραστηριότητες που δυσκολεύουν αφάνταστα την καθημερινή τους ζωή. Και έχουμε δει μητέρες που, που μαθαίνουν τα παιδιά τους να πίνουν γουλιά γουλιά το νερό διότι άμα τελειώσει η ταμιτζάνα ας πούμε ε, θα πρέπει να ξαναπερπατήσουν όλα αυτά τα χιλιόμετρα να πάρουν πόσιμο νερό. Αυτά τα προβλήματα αυξάνονται συνέχεια στις παράκτιες περιοχές και όλο και περισσότερο εκατομμύρια αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του νερού που δεν είναι πόσιμο, επειδή είναι υφάλμηρο. Επίσης πάρα πολλοί κάτοικοι δυσκολεύονται ιδιαίτερα να καλλιεργήσουν ε, ε, καλλιέργειες οι οποίες είναι εποφελείς οικονομικά. Αναγκάζονται ή να καλλιεργούν ε, ρύζι, τροφές οι οποίες είναι λιγότερο αποδοτικές οικονομικά ή να μετικούν, να φύγουν, να εγκαταλείψουν τη γη τους, τα χωράφια τους και να οδεύσουν προς τις πόλεις, προς τις αστικές περιοχές. Στις νότιες περιοχές του Μπαγκλαντές τα τελευταία 20 χρόνια δεν, έχει, δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές δημογραφικές τα δημογραφικά στοιχεία όμως μας δείχνουν ότι ο αριθμός των γυναικών και των παιδιών αυξάνεται, ενώ ο αριθμός των ενήλικων ανδρών μειώνεται, που σημαίνει ότι δεν έχουν αλλάξει σημαντικά οι αριθμοί του, τα στοιχεία, τα σημαντικά στοιχεία του πληθυσμού, αλλά φεύγουν οι ενήλικες άντρες από τις παράλιες περιοχές, παράκτης περιοχές και, και μεταναστεύουν προς τις αστικές περιοχές. Αυτές είναι λίγες από τις σοβαρές επιπτώσεις τις οποίες έχουμε σημειώσει τα τελευταία χρόνια και που σχετίζονται άμεση με την κλιματική αλλαγή. Η Πρόεδρος, θα δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή, στην Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τον Παγκλαντές. Ε, μερικούς τους γνωρίζω πολύ καλά από τις διαπραγματεύσεις και χαίρομαι πολύ που τους ξανασυναντώ εδώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσίασή σας ε, και για την παρουσία σας εδώ. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπετε την ευρύτερη εικόνα ε, πριν από μας ε, και εν ώψη των διαπραγματεύσεων και στη Βασοβία αλλά και πιο μετά στο Παρίσι. Υπάρχει προσαρμογή που είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως επίσης και το θέμα της άμβλυνσης γιατί αν δεν αμβληνθούν οι προσπάθειες προσαρμογής ε, θα είναι πολύ πιο δαπανηρές στο μέλλον και μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η προσαρμογή αυτή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και οι δύο πτυχές, προσαρμογή και άμβληση, να θεωρηθούν ως τμήμα ε, του ίδιου πράγματος και όχι αντιφατικές, γιατί μερικές φορές τι ε, διαπραγματεύσεις δημιουργούνται δημιουργείται κατά λάθο μια αντίφαση μεταξύ των δύο και πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δύο ζητήματα από κοινού. Τώρα όσον αφορά τη χρηματοδότηση για την προσαρμογή, όπως είπατε είναι πολύ σημαντικό να τη συμπεριλάβουμε στην αναπτυξιακή βοήθεια και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούμε είναι απολύτως απαραίτητο να την συμπεριλάβουμε για να εξασφαλίσουμε ότι οι αναπτυξιακές προσπάθειες ε, είναι βιώσιμες και δεν θα ε, χαθούν λόγω των κλιματικών αλλαγών. Από την πλευρά λοιπόν του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 400 εκατομμύρια ευρώ ε, ε, δόθηκαν από το 2007 ως το 2013 για τον Μπαγκλαντές, 30 εκατομμύρια σε καταπίστευμα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για τους πιο φτωχούς και για τους πιο ευάλωτους το 2011 και εκτός από αυτό Έχουμε δουλέψει πολύ για την επισητιστική ασφάλεια και για άλλα ζητήματα στον Παγκλαντές, τα οποία έχουν άμεση σχέση με το θέμα της προσαρμογής αλλά και της άμβλυνσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό τα στοιχεία, τα, τα, τις πτυχές του κλίματος να τις, συμπεριλάβουμε, να τις συμπεριλάβουμε στην αναπτυξιακή μας συνεργασία. Όσον αφορά την κινητοποίηση κονδυλίων από τις θεματικές μας ε, γραμμές, για παράδειγμα υπό τη Συμμαχία ε, για την αλλαγή ε, του κλίματος, 8,5 εκατομμύρια το 2009, όπως επίσης και επισητιστική βοήθεια το 2007, 36,8 εκατομμύρια και το 2012 άλλα 18 εκατομμύρια. Οπότε υπάρχουν μεγάλα ποσά που έχουν δοθεί και είναι δημόσιες, ε, ε, δημόσιες ε, επιδοτήσεις προς τον Παγκλαντές. Συμφωνούμε ότι χρειάζεται την υποστήριξη αυτή των Παγκλαντές και θα συνεχίσουμε να το βοηθάμε. Ακόμα και στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχουμε ακόμη οικονομικά νούμερα γιατί υπάρχουν ακόμη διαπραγματεύσεις για τα σχετικά νομικά μέσα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αλλά μπορούμε να πούμε ότι θα συνεχίσει η υποστήριξη του, του Μπαγκλαντές. Να περάσω τώρα στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής σας που είναι η άμβλυνση η προσπάθεια άμβλυνσης των ε, συνεπειών. Χωρίς αυτές τις προσπάθειες η προσαρμογή θα είναι πάρα πολύ δαπανηρή στο μέλλον. Είναι απλά τα πράγματα. Αν θέλουμε να μείνει κάτω από δύο βαθμούς ε, η παγκόσμια θέρμανση ε, του κλίματος, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Η Βασοβία ε, πρέπει να είναι η βάση για αυτή την ενισχυμένη συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πρόθεση να κάνει περισσότερα. Έχουμε μονομερώς υποβέλει έναν στόχο μείωσης κατά 20% μέχρι το 2020 και ε, προσπαθούμε να ε, ενισχύσουμε τους στόχους μας για το 2030, να έχουμε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους το 2030. Τώρα, πώς, πόσο φιλόδοξο μπορεί να είναι αυτό ο στόχο, αυτό εξαρτάται από τι διεθνεί διαπραγματεύσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει ηγεσία να πρωτοστατήσει σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τη δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Αυτή τη στιγμή οι εκπομπέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 10 με 11% των παγκοσμίων εκπομπών. Αυτό σημαίνει ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει τι εκπομπέ και οι υπόλοιποι όχι, δεν θα επιτύχουμε. Πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε και αυτή η, η νέα συμφωνία αποτελεί μία ενορχίστρωση όλων αυτών των προσπαθειών ε, γιατί όλοι πρέπει και να υποσχόμαστε αλλά να μπορούμε να αναλαμβάνουμε και το δικό μας τμήμα της ευθύνης. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε μεν τους, ε, τις φιλοδοξίες μας αλλά να έχουμε και μία νομική δεσμευτική συμφωνία, δεσμευτική συμφωνία το 2015. Είναι σημαντικό για να γίνει αυτό τα μέρη που ενδιαφέρονται περισσότερο, οι πιο ευάλωτες, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, να δεσμευθούν και εκείνες, ε, να συνεργαστούν με ανεπτυγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες χώρες ε, που θέλουν να δουν μια τέτοια νομικά δεσμευτική συμφωνία να ισχύει και όλοι να λειτουργήσουν στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Τώρα τι μπορούμε να επιτύχουμε στη Βαρσοβία. Έχουμε μάθει από το παρελθόν και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην φτάνουμε μέχρι τον τελευταίο μήνα πριν από την, τελευταία, από την τελική συμφωνία. Ήδη από το 2014 νομίζω ότι πρέπει να δράσουμε. Είναι η στιγμή για όλα τα μέρη να ε, δώσουν υποσχέσεις άμβλυνσης και πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτές στην πράξη, σε ποιο βαθμό είναι συγκρίσιμες και σε ποιο βαθμό μας επιτρέπουν να επιτύχουμε τους στόχους μας, δηλαδή τη διατήρηση της παγκόσμιας θέρμανσης κάτω από δύο βαθμούς. Νομίζουμε ότι αυτό θα ήταν μια καλή ε, έκβαση της Βαρσοβίας, αν έχουμε κάποια κοινή μορφή των υποσχέσεων αυτών, πληροφορίες που θα έπρεπε όλα τα μέρη να υποβάλουν ε, σε σχέση με τις προτινόμενες δεσμεύσεις. Είναι πάρα πολύ τεχνικά αυτά, αλλά είναι σημαντικό να προοδεύσουμε για το θέμα των λογιστικών κανόνων που τις συνοδεύουν ε, τις υποσχέσεις αυτές για να ξέρουμε τι ακριβώς θα πει όταν έχουμε μειώσει τις εκπομπές, ότι ένας τόνος μείωση στην Ευρώπη είναι ίδιος με τον ένα τόνο στις ΗΠΑ ή στην ε, Ασία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα ε, της ε, νέας συμφωνίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ο Μπαν Κιμούν, είπε ότι θέλει να δει τα μέλη να υποβάλουν συγκεκριμένες υποσχέσεις μέχρι του χρόνου και τότε οι, οι ηγέτες όλου του κόσμου το Σεπτέμβριο του 2014 θα συνέλθουν για να ε, το συζητήσουν και ε, εφόσον θα είναι διαθέσιμες αυτές οι υποσχέσεις ε, θα μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη όθηση στις διαπραγματεύσεις και να φτάσουμε στο είδος αυτό της συμφωνίας που χρειαζόμαστε. Υπάρχει λοιπόν κάποια όθηση και βασιζόμαστε στην βοήθεια του Μπαγκλαντές και άλλων αναπτυσσομένων χωρών Λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να ολοκληρώσω κάπου εδώ. Ευχαρίστω ε, να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, καλεσμένους μας από το Μπαγκλαντές για τις ε, ομιλίες τους, για τις προφορίες που μας έδωσαν και για την υποστήριξη που έδειξαν προς ε, τη συνεργασία μας και όλες τις συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ μας. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή και σας διαβεβαιώ ότι έχουμε απόλυτη δέσμευση προς τους κοινούς μας στόχους. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε για λίγα λεπτά να προσέλθει ο πρόεδρος του Πράσινου Κροτήριου, ο οποίος έχει τώρα εισέλθει στην αίθουσα. Ε. Can I just add... Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάτι πολύ σύντομα για το τι κάνουμε στο Μπαγκλαντές. Είμαι από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, στην Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή προετοιμάσουμε το επόμενο πρόγραμμα βοήθειας για τα επόμενα 7 χρόνια και επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε τρεις τομείς, τρεις τομείς μόνο. Και βεβαίως ε, ε, ένας από τους τρεις αυτούς τομείς είναι η ασφάλεια τροφίμων και, και τα τρία αυτά και τρεις αυτές πτυχές συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Έχουμε λοιπόν τρία προγράμματα για τα επόμενα 7 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα υποδεχτούμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση τον ε, κύριο Ζόρζ Κάρλος Φονσέκα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακροτηρίου. Θα ανταλλάξουμε απόψει μαζί του σχετικά με τι κοινωνικέ και οικονομικέ εξελίξει του Πράσινου Ακροτηρίου και τη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημοκρατική σταθερότητα του Πράσινου Ακροτηρίου και η ποιότητα τη κυβέρνησή του, που έχουν αποδειχθεί από του δείκτε ε, που παρουσίασαν ε, οι διεθνείς οργανώσεις δώνουν ε, την εικόνα μιας χώρας μοντέλου για πολλές άλλες ε, χώρες αναπτυσσόμενες. Το γεγονός ότι είστε μεταξύ των χωρών που έχουν καταφέρει να πετύχουν τους στόχους της ηλετίας που θα καταφέρουν μάλλον να πετύχουν του στόχου λήπτη το 2015 είναι αξιοσημεία. Το Πράσινο κροτήρι, επίση είναι μία από τι σπάνιε χώρε που βγήκε από τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε, από την ομάδα αυτή των χωρών. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν να είναι υψηλέ οι κοινωνικέ ανισότητε, έχει αυξηθεί η ανεργία και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα σε σχέση με την κατάσταση των γυναικών. Η σχέση σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρή και αντικατοπτρίζει τα πολλά κοινά μας ενδιαφέροντα. Η επιτυχία της χώρας σας στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί παράδειγμα. Μεταξύ των πολλών θεμάτων που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι και αυτό που συζητήσαμε με τους εκπροσώπους από τον Μπαγκλαντές, ε, την κλιματική αλλαγή. Αυτό μας αφορά όλους ε, και ε, τις ε, χώρες, τις άγονες, τις περιοχές του Σαχέλ αλλά και το πράσινο κροτήρι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή. Χαιρόμαστε πολύ που σας υποδεχόμαστε εδώ κύριε Πρόεδρε για να συζητήσουμε ακριβώς τα θέματα αυτά. Πριν να σας δώσω το λόγο, ο συνάδελφος, ο κύριος Μπρόκ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, θα κάνει μια σύντομη εισαγωγή. Είμαστε πράγματι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που γίνεται αυτή η κοινή συνεδρίαση μεταξύ των δύο επιτροπών μας. Κύριε Μπρόκ. Κυρία Ζολή, κύριε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με πολύ εξαιρετική χαρά Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά σα υποδέχομαι σήμερα εκ μέρου της επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Όπως είπε και η Πρόεδρος μας, κυρία Ζολή, η χώρα σας έχει σημειώσει ε, μεγάλη επιτυχία. Είναι μια χώρα επιτυχίας. Ε, έχει μια σταθερή δημοκρατία, ένα υπόδειγμα καλής διακυβέρνησης και πιστεύω ότι αυτό είναι λίγαν εντυπωσιακό. Ε, έχετε προοδεύσει και έχετε γίνει μια χώρα μεσαίων εισοδημάτων και είσαστε καθοδόν προς την επίτευξη των στόχων της ε, χιλιετίας στο 2015. Μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας Θεωρήσεων και Επανεισδοχής πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει ακόμα περισσότερο διότι μας δίνεται δυνατότητα όχι μόνο να ε, συστήξουμε περισσότερο τις σχέσεις μας, αλλά να ενισχύσουμε και την ανάπτυξη και τη διμερή συνεργασία. Με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να δώσουμε ένα νέο έναυσμα ε, στις σχέσεις μας και να εργαστούμε ε, μαζί για την επίτευξη των στόχων μας που βασίζονται στις κοινέ μας αρχές. Ε, αντιμετωπίζουμε πολλές μεγάλες προκλήσεις. Από ε, πλευράς Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων γνωρίζουμε και τα προβλήματα που έχετε με τα, με διακίνηση ναρκωτικών, με τη βία, με απειλές από την ευρύτερη περιοχή και βεβαίως θα μας, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μάθουμε πώς ε, προβλέπετε να επιτύχετε περαιτέρω πρόοδο για την, ε, πρόοδο, συγγνώμη, για την καταπολέμηση αυτών των σοβαρών προβλημάτων, την καταπολέμηση για ναρκωτικών, βίας και, και επίσης με την η συνεργασία με την ΕΚΟΒΑΣ θα καταλήξει στην επικύρωση της ε, σύμβασης που θα αποτελέσει άλλο στοιχείο επιτυχίας για τη χώρα σας. Πιστεύω ότι η χώρα σας μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα σχέσεων με άλλες χώρες και αμοιβαία υποστήριξης και βοήθειας. Ε, χαίρομαι, επαναλαμβάνω και πάλι που βρίσκεστε εδώ μαζί μας και σας δίνω το λόγο. Muito tarde. Καλησπέρα σε όλους. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Ανάπτυξης, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι Υπουργοί Εξωτερικών του Πρασινοκριτηρίου, κυρίες και κύριοι δημοσιογράφοι, ως ε, πρόεδρος ε, της Δημοκρατίας ε, και ως ύπατος εκπρόσωπος του έθνους μου παρουσιάζω τους χαιρετισμού όλων των συμπατριώτων μου, των συμπατριωτών μου που ζουν και στα νησιά αλλά και στις κοινότητες του εξωτερικού και κυρίως όσων ζουν στην Ευρώπη. Δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά την πρόσκληση που μου υπευθύνθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς και Είμαι εδώ ενώπιόν σας, ενώπιον των εξοχότητών σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε μια κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών εξωτερικών υποθέσεων και ανάπτυξης. Θα εκμεταλλευτώ αυτά τα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου για να σας γνωστοποιήσω πώς ερμηνεύουμε εμείς τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός ε, και την πολιτική, οικονομική και κοινωνική διαδρομή της χώρας μου, του Πράσινου Ακροτηρίου. Το Πράσινο Ακροτήρι είναι ένα μικρό νησιωτικό κράτος, ε, ε, βρίσκεται στο αρχιπέλαγος της ακτής της Δυτικής Αφρικής. Ε, γνωρίζετε ότι δεν έχει τους παραδοσιακούς πόρους. Ε, οι κλιματικές συνθήκες ε, είναι δύσκολες και οι άνθρωποι, οι άνδρες και οι γυναίκες στη χώρα μου αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις και προσπαθούν να αποτελέσουν μια προηγμένη δημοκρατία, να δημιουργήσουν μια χώρα ανταγωνιστική και αναπτυγμένη. Πέραν των πολλών δυσκολιών στα 38 χρόνια της ανεξαρτησίας μας και στα πάνω από 20 χρόνια δημοκρατίας νομίζω ότι το πράσινο κροτήρι αποτελεί πλέον ένα κράτος δικαίου και είναι ένα ενεργό μέλος διάφορων διεθνών οργανώσεων, Αφρικανικής Ένωσης, ε, του, των Ηνωμένων Εθνών ε, και των, ε, χωρών, των πορτογαλόφωνων χωρών, της κοινότητας των πορτογαλόφωνων χωρών. Συμμετέχει στη διεθνή κοινότητα με διμερείς αλλά και πολυμερείς σχέσεις και φυσικά έχουμε και μία ιδιαίτερη σχέση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία εταιρική σχέση από το 2007. Εμείς ε, κερδίσαμε την εξαρτησία μας το 1975 με πολύ δυσίωνες προοπτικές. Ε, ξεκινούσαμε από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ε, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι κάποιοι έλεγαν ότι δεν θα είναι βιώσιμο το μέλλον μας, όμως εμείς καταφέραμε να οικοδομήσουμε μια χώρα, να οικοδομήσουμε ένα κράτος και σήμερα βιώνουμε μία προηγμένη και σύγχρονη δημοκρατία. Η διαδρομή του πρασινοκροτηρίου ήταν ευτυχώς ειρηνική και σταθερή και όλοι το λένε ότι ήταν καλή η διακυβέρνηση και είχαμε ένα όραμα για την πρόοδο και ε, καταφέραμε με αυτόν τον ε, τρόπο να αυξήσουμε το κατακεφαλή εισόδημα και έτσι το πράσινο ακροτήρι κατόρθωσε να βγει από την ομάδα των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Όταν ε, ε, κερδίσαμε την ανεξαρτησία μας, είχαμε ένα κατακεφαλή ΑΕΠ 129 αμερικανικών δολαρίων, ενώ τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 3.000 αμερικανικά δολάρια. Και εκμεταλλευτήκαμε ε, αυτή την αύξηση του ΑΕΠ ως ένα παράθυρο ευκαιρίας για σύναψη εταιρικών σχέσεων και μέσω της συνεργασίας θα μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις ε, σε νέες απαιτήσεις ε, της σημερινής διαδικασίας ανάπτυξης. Αναφέρομαι στην ατότητα και ενεργοποίηση, σε καινοτόμου χρηματοδότηση σε άμεσε ξένες επενδύσει και σε άλλες ε, μορφές εταιρικών σχέσεων και επενδύσεων που μπορούν να αφαιρούν και τα δύο μέρη. Στη βάση αυτή δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε ε, κάποιες δικαιολογίες ε, για να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη του πράσινου κροτηρίου πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε σήμερα στον ε, ε, πρόεδρο Μπαρόσο ότι για μας η προσπάθεια που έχει γίνει για να αναβαθμιστούμε, δηλαδή για να περάσουμε από μια λιγότερο αναπτυγμένη χώρα σε μια χώρα με μέσο εισόδημα, όλη αυτή, όλη η προσπάθεια να οικοδομήσουμε ένα κράτος δικαίου, να είμαστε μια χώρα που σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπου ο βαθμός ε, ανοχής είναι μεγάλος ε, και από την ε, στιγμή της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας είδαμε πολλές εναλλαγές και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την αναλλαγή της εξουσίας και αυτό πάντοτε υπό κανονικές συνθήκες. Και εγώ ως πρόεδρος της Δημοκρατίας του Πράσινου Συνοκροτηρίου εδώ που μόλις έχω εγώ δύο χρόνια ε, θητεία ε, εξελέχθη και έξι μήνες μετά από τις εκλογές ε, όπου νίκησε ένα κόμμα που δημιούργησε. Ε, μια ανακυβέρνηση. Εγώ εκλέχτηκα όμως δεύτερη φορά χωρίς την υποστήριξη του κυβερνητικού κόμματος. Έτσι λοιπόν, με τη δική μου εκλεγή, το πράσινο ακροτήρι αυτή τη στιγμή βιώνει μια νέα δημοκρατική εμπειρία. Δηλαδή έχει ένα πρόεδρο της δημοκρατίας, ο οποίος δεν προέρχεται από την ίδια πολιτική οικογένεια ε, με το κόμμα που κυβερνά αυτή τη στιγμή. Και παρόλα αυτά λειτουργούμε με σταθερότητα, χωρίς να προκαλείται κανένα είδος κρίσης. Και θα σας πω ότι σε 22 χρόνια δημοκρατίας ποτέ στη χώρα μου δεν υπήρξε κάποια πολιτική κρίση. Είχαμε τα συνήθη προβλήματα δημοκρατικής δυναμικής, αλλά πάντοτε επιλύονταν ε, μέσα στο θεσμικό πλαίσιο και φυσικά στο πλαίσιο του συντάγματος ε, του 1992. Ποτέ δεν είχαμε πρόορες εκλογές από το 1992 Έχουμε υλοποιήσει έξι ε, εκλογές ε, τοπικής αυτοδιοίκησης και τέσσερις νομοθετικές, βουλευτικές εκλογές. Ή πέντε. Και πέντε προεδρικές εκλογές και όλοι έφτασαν μέχρι το τέλος της θητείας. Και πρόκειται αντικειμενικά για μία μοναδική περίπτωση τουλάχιστον ε, αν λάβετε υπόψη την ευρύτερη περιοχή, την Αφρική. Αν ε, εμείς λοιπόν αναβαθριστήκαμε σε χώρα αμέσως εισοδήματο και αν όλοι εδώ μας, δίνετε κίνητρα βάση δημοκρατικών εμπειριών και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτή η αναβάθμιση πρέπει να αποτελέσει ένα στοιχείο υποστήριξης και περαιτέρω συνεργασίας, περαιτέρω κινήτρων. Δεν μπορεί να αποτελεί ένα μειονέκτημα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο εμείς πάντοτε υπερασπίζουμε τους εαυτούς μας και σήμερα ακούμε ενθαρρυντικά λόγια. Ελπίζουμε ότι και οι ευρωβουλευτές που παρευρίσκονται εδώ θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι στα πλαίσια του 21ου ε, φέτο ο φάκελος ε, για το πράσινο κροτήρι δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο, στο κορδίλι δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από τα προηγούμενα έτη. Και πρέπει να δοθούν περαιτέρω κινητρά στη χώρα μας για να σημειώσει πρόοδο, για να μεταφράσει και στην πράξη αξίες που είναι κοινέ για όλους μας. κύριε κύριοι πρόεδροι και αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, για μένα, για μας, το θεμέλιο της ειδική εταιρικής σχέσης, ε, το κύριο στοιχείο της ιδιαίτερης σχέσης που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να είναι η δυνατο... το ότι εμείς συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες, ότι πιστεύουμε στην ελευθερία, ότι πιστεύουμε στη δημοκρατία, ότι πιστεύουμε στο κράτος δικαίου στην ανοχή, στο σεβασμό της διαφοράς. Στο ότι πιστεύουμε στο διάλογο, στη διπλωματία για την επίλυση των σειράξεων μεταξύ των εθνών και των λαών. Εμείς είμαστε μια χώρα πολιτικά και κοινωνικά σταθερή και αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε ένα πολιτισμό ανοχής ε, και κοινών αξιών. Και γι' αυτό εμείς θεωρούμε πως η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε καμία ψευδέστηση. Δεν ε, θεωρούμε τον εαυτό μας ε, μία ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, είμαστε μια χώρα με ιδιαιτερότητες. Όμως θέλουμε να εργαστούμε και ονειρευόμαστε αυτή η σχέση να ενισχυθεί και εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε και μέχρι το όριο του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να βρούμε και νέα μέσα συνεργασίας που αποτελούν, θα αποτελούν συνιστώσεις της σταθερότητας. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών, να υπάρχει τεχνική και κανονιστική σύγκληση και αυτά που είπατε προηγουμένως, ε, κυρία Πρόεδρε, θέλουμε να μειώσουμε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής σε χώρες νησιωτικές όπως είναι το πράσινο ακροτήρι. Και φυσικά αυτό στα πλαίσια της προοπτικής να χρησιμοποιήσουμε και τις ενενεώσιμες πηγές ενέργειας, να προστατεύσουμε περισσότερο το περιβάλλον, να δημιουργήσουμε μια οικονομία που θα είναι και πράσινη αλλά και γαλάζια. Και πάντοτε μιλάμε για εξέλιξη εμείς, γιατί πρόκειται για, για εμείς ξεκινήσαμε από μια συμφωνία που βασιζόταν ε, στο Κοτονού, αλλά φτάσαμε σε αυτή την ειδική εταιρική σχέση και μπορέσαμε να αναπτύξουμε τους πυλώνες της σχέσης αυτής. Και εγώ εδώ θα ολοκλήρωνα την παρέμβασή μου, για να μην μακρηγορήσω, λέγοντάς σας ότι εμείς δεν έχουμε μια τέλεια δημοκρατία, δεν ξέρω καν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανεπάρκειες και ελλείψεις στο κράτος δικαίου μας. Πολλές ε, φορές ε, και εγώ ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρομαι στον αδύναμο χαρακτήρα του σημερινού κράτους δικαίου. Εγώ έχω πει παραδείγματος χάρη ότι στο πράσινο κρατήρι δεν έχουμε ακόμη μια τόσο διευρυμένη δημοκρατική κουλτούρα, μια τόσο ισχυρή δημοκρατική κουλτούρα όπως τα ονειρευόμασταν. Ίσως δεν έχουμε ακόμη και ένα δικαστικό σύστημα που από τεχνική σκοπιά να λειτουργεί όπως πρέπει. Δεν έχουμε ακόμη στο πράσινο ακροτήρι μια ισχυρή κοινή γνώμη μία κοινή γνώμη που να λειτουργεί ως ένα τύπο δικαστήριο κατά κάποιο τρόπο ελέγχου όλων των εξουσιών. Δεν το έχουμε αυτό στη χώρα μου. Ούτε βρισκόμαστε σε μια ηγετική θέση, παρόλο που όταν παραδείγματος χάρη μια πρόσφατη, όταν μια πρόσφατη έκθεση θεώρησε ότι είμαστε η 26η δημοκρατία του κόσμου. Τότε αισθανθήκαμε μεγάλη περηφάνεια. Όμως ε, δεν το κάναμε εμείς αυτό τον κατάλογο, δεν το καταρτήσαμε εμείς και αυτό μας έκανε περήφανους. Αλλά όλα αυτά κυρίως μας έδωσαν κίνητρα για να έχουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, για να καταστήσουμε ανταγωνιστική τη χώρα μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον οικονομικής ανταγωνιστικότητας, γιατί στο πράσινο κροτήρι ξέρουμε ότι ο καιρός ε, των ε, δανείων, ε, των εκχωρήσεων φτάνει στο τέλος του και πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εσωτερικές συνθήκες για να καταστήσουν ανταγωνιστική την οικονομία. Να δημιουργήσουμε μία μικρή οικονομία υπηρεσιών. Για να σας δώσω μία ιδέα, αυτή τη στιγμή στο πράσινο κροτήριο τουρισμός, αν σκεφτούμε μόνο τα άμεσα έσοδα, φτάνει περίπου στο 22-23% του έκπατς. Και αν ε, βάλουμε και τα έμεσα έσοδα, ο τουρισμός σήμερα μπορεί να φτάνει πάνω από το 45% της χρηματοδότησης της οικονομίας μας. Αλλά μια τέτοια οικονομία επηρεάζεται από τις συνθήκες ε, και επηρεάζεται από τον αντίκτυπο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η δική μας οικονομία ήταν εξαρτημένη από την οικονομία των χωρών του ευρώ μέχρι σήμερα και γι' αυτό εμείς καταβάλουμε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσουμε την οικονομία μας, αλλά επίσης συνειδητοποιούμε και άλλα προβλήματα που ανέφερε εδώ ο Πρόεδρος το θέμα της εγκληματικότητας, της, του οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος. Στο πράσινο ακροτήρι και λόγω της γεωγραφικής μας θέσης η χώρα μας έχει χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για τη διακίνηση ναρκωτικών και για, για τη διακίνηση άλλων προϊόντων. Ο διάδρομος του Ατλαντικού ήταν στόχος ε, της ε, επιχείρησης θαλάσσιας όλες. Εμείς δεν είμαστε μακριά από τον κόλπο τη Γουινέα, όπου η πειρατεία, η θαλάσσια πειρατεία είναι ένα σοβαρό φαινόμενο. Ξέρουμε ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών και σε γειτονικέ χώρε. Αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι και βάσει του ρόλου που έχω εγώ στο σύστημα κυβέρνησης ε, της ε, χώρας μου ως πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορώ να σας πω ότι θεσμοί στο πράσινο ακροτήρι οι αστυνομικές αρχές, οι διοκτικές αρχές έχουν κάνει μία αξιοσημείωτη προσπάθεια για να καταπολεμήσουν αυτά τα φαινόμενα. Αρκεί να πούμε ως παράδειγμα όταν ε, εγώ ε, υλοποιώ αυτή την επίσκεψη στην Ευρώπη, μου γνωστοποιήθηκε η, ε, η κατάσχεση μιας σημαντικής ποσότητας ε, κοκαίνης από τις αστυνομικές μας αρχές με συνεργασία και με δυνάμεις άλλων χωρών. Έχουμε συνεργαστεί με την Ισπανία, με τη Γαλλία, με τη Βραζιλία, με τις Ηνωμένε Πολιτείε, με την Πορτογαλία σε θέματα καταπολέμησης διακίνησης ναρκωτικών. Όμως δεν μπορούμε να δώσουμε μόνοι μας αυτή τη μάχη, δεν διαθέτουμε τα μέσα, δεν έχουμε την ικανότητα να δώσουμε αυτή τη μάχη χωρίς διάρθρωση με τις άλλες χώρες, ούτε χωρίς στήριξη από τη διεθνή κοινότητα, αλλά έχουμε αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις και δίνουμε αποφασιστική μάχη κατά της διακήρυξης ναρκωτικών και του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος η Γενική Εισαγγελία έχει υλοποιήσει μια γενικευμένη δράση για να τελειοποιήσει την καταπολέμηση της νομοποίησης παρανομοσόδων. Είναι πρόβλημα που έχουμε. ξέρετε ότι εμεί είχαμε ένα πρόβλημα με το χρηματιστήριο. Ο διευθυντής ε, του χρηματιστηρίου είναι υποκράτηση αυτή τη στιγμή. Δεν ε, έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δικαστική διαδικασία ε, και δεν μπορούμε λοιπόν να τοποθετηθούμε για το θέμα αυτό. Όμω όλα αυτά μας δείχνουν ότι λειτουργούν οι θεσμοί στο πράσινο κροτήρι και ότι δίνουμε αυτή τη μάχη, αυτό τον αγώνα. Τώρα, σε σχέση με την οικονομική συνεργασία με τον ΟΣΑ. Εμείς ε, θέλουμε να είμαστε ένας χρήσιμο εταίρος. Ε, εμείς έχουμε κατανοήσει ότι δεν θέλουμε να είμαστε απ' έξω, θέλουμε να είμαστε ένας πλήρης εταίρος και να συμμετέχουμε ε, σε οργανώσεις όπως ε, είναι η Αφρικανική Ένωση, οργανισμοί που προωθούν την ε, δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως δυστυχώς Είχε δημιουργηθεί στην αρχή μια Οικονομική Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, στα, ε, στα πλαίσια της ΕΝΤΕΟ και πάρα πολλές συγκρούσεις ε, έλαβαν χώρα. Ξέρετε την περίπτωση του Μαλή, της Γουινέας Μπισάου και άλλες χώρες της, που ανήκουν στη ΣΕΝΤΕΟ. και πολλά από τα κονδυλία και τις προσπάθειες του χρησιμοποιούνται για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Εμείς ελπίζουμε τελικά η ΣΔΕΟ να μπορέσει πραγματικά να ασχοληθεί με θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και οικονομικής ανάπτυξης των χωρών που συμμετέχουν στην κοινότητα αυτή. Και για να κλείσω, θα ήθελα μια ακόμη φορά, εξ ονόματος ολόκληρου του λαού μου, να σας ευχαριστήσω για την ένθερμη υποδοχή σας. Και θα ήθελα ιδίως να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Αντιπρόεδρο και τους Πρόεδρους των Επιτροπών που μας υποδέχτηκαν και επίση να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεισφορά του στην ε, μόνιμη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πράσινου Κριτηρίου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές. Πρώτα ο κύριος Γκέρενς. Χρόνος ομιλίας 4 ε, λεπτά για κάθε ευρωβουλευτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τον πρόεδρο του Πράσινου Ακροτηρίου. Εδώ είμαι. Είπατε ότι είναι, είστε μια ιδιαίτερη χώρα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια χώρα όχι σαν τις υπόλοιπες και δεν το λέω με αρνητική χρειά. Δεν πρέπει να το πάρετε άσχημα. Το εννοώ αντιθέτως ως κομπλιμέντο. Θυμάμαι την πετάβαση της χώρας σας ε, από το καθοστέως ε, της λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας ε, σε μια ενδιάμεση χώρα και όλο το δράμα της, του διαλόγου στο πράσινο ακροτήρι για την χρήση της βοήθειας οποίας, ε, ε, της οποίας ήσασταν δικαιούχος. Ε, η μετάβαση αυτή, κατά τη γνώμη σας, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Οπότε, μου γεννιέται το εξής ερώτημα. Η σχέση μεταξύ της χώρας σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Η εταιρική μας σχέση. Η αναπτυξιακή συνεργασία είναι η βασική πτυχή της συνεργασίας αυτής εκτός από τις πολιτικές σχέσεις στις οποίες αναφερθήκατε αλλά νομίζω ότι υπάρχουν δύο δυνατότητες. Η μία ε, είναι η συνέχιση αυτής της μετάβασης ε, που σας έχει, έχει δώσει τη δυνατότητα να σημειώσετε πολύ σημαντικό, σημαντική πρόοδο και στον εκδημοκρατισμό αλλά και ε, από απόψεις οικονομικής ανάπτυξης. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι υπήρχε στην Κρουσέντ μία έκθεση το ευάλωτον της πράσινη, του πράσινου ακροτηρίου. Ε, πάντοτε λοιπόν η χώρα σας ε, ήταν ευάλωτη σε πράγματα τα οποία δεν μπορείτε πάντοτε να χειριστεί, ε, η επιτηρητιστική εξάρτηση της χώρας σας, η κλιματική αλλαγή, όπως επίσης και τότε η εξάρτηση της χώρας σας... Ε, ε η μεγάλη διασπορά ε, κονδυλίων ε, της οποίας, των οποίων ήσασταν δικαιούχοι. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και είναι ένα ερώτημα το οποίο απευθύνω και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πάρα πολύ σημαντικό από πολιτικής απόψεως. Ε, αυτή τη στιγμή αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για το, τους στόχους του 2020 όπως επίσης και στο ε, ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, αναρωτιόμαστε σε σχέση με το μέλλον των συνεργατών μας των συνεταίρων μας για παράδειγμα συμφωνίες όπως για παράδειγμα με τις Κανάριες νήσους ε, Συμφωνίες Interreg. Μήπως θα μπορούσαμε λοιπόν, ε, θα μπορούσαμε και υπό άλλες μορφές να δούμε τη συνέχιση αυτής της μετάβασης μέσω του Interreg για παράδειγμα. Ε, ένα παράδειγμα δίνω. γιατί κι εσείς ε, λέτε ότι έχετε ένα ιδιαίτερο καθεστώς στη σχέση σας με ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η κυρία Καβάγιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τιμή μας είναι να σας πω ότι είμαστε εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε. Το Πράσινο Κρατήριο αποτελεί ένα καλό παράδειγμα καλής διακυβέρνησης, δημοκρατίας και καλής χρησιμοποίησης της ε, αναπτυξίας βοήθειας. Αυτές οι πτυχές ε, έδωσαν τη δυνατότητα στο πράσινο κροτήρι να έχει μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το πράσινο κροτήρι είναι μια χώρα ε, μεσαίας ανάπτυξης και εγώ ε, ως ε, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, και Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, έχω πει ότι δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί το πράσινο κροτήρι λόγω αυτής της αναβαθμίσης του. Το αντίθετο, πολλοί ευρωβουλευτές όταν εκπονούν τις διάφορες εκθέσεις τους έχουν κατά νου το τι συμβαίνει στο πράσινο κροτήρι. Παραδειγματικά θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, εισήγηση της κυρίας Γκόμπες σε σχέση με ε, την θαλάσσια πολιτική και ασφάλεια ε, και άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Γκόμες, δεν βρίσκεται εδώ σήμερα, αλλά μου ζήτησε να φερθώ συγκεκριμένα στην έκθεσή της, η οποία υπογραμμίζει το στρατηγικό ρόλο του πράσινου κροτηρίου στην ασφαλή του Ατλαντικού. Όμως, αυτή ε, ε, πρόκειται ε, ουσιαστικά κάτι που το βρίσκουμε συνεχώς στις εκθέσεις των διάφορων συναδέλφων για θέματα ενέργειας, ασφάλειας, αλίας. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να είστε σίγουρος ότι έχετε πάρα πολλούς φίλους της χώρας σας εδώ. Όπως και εσείς είπατε, η ειδική εταιρική σχέση θα διευκολύνει νέες επενδύσεις σε καινοτόμους τομείς. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στους τομείς με τους οποίους ασχολούμαι περισσότερο και που πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία για το πράσινο ακροτήρι σε αυτή την νέα εποχή συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να αναφερθώ στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην ανώτατη εκπαίδευση και ξέρω ότι γίνεται πολύ λόγος ε, για την ε, ανώτατη εκπαίδευση στο πράσινο κριτήριο γιατί δημιουργήθηκε και με τη βοήθεια της ε, Πορτογαλίας ένα ε, δημόσιο πανεπιστήμιο στη χώρα σας και φυσικά αυτό μπορεί να βοηθήσει στην κινητικότητα των φοιτητών και των ερευνητών. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και στις καινοτόμες, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Θα ήθελα να σας ζητήσω ένα σχόλιο για αυτό το νέο κύμα νέων πολιτικών συνεργασίας. Πώς εσείς βλέπετε το ρόλο των ευρωβουλευτών. Πώς μπορούμε εμείς να διευκολύνουμε οι χώρες σας και οι θεσμοί σας να μπουν σε αυτά τα δίκτυα, σε αυτές τις εταιρικές σχέσεις με πανεπιστήμια, με μικρές και μεσές επιχειρήσεις των διαφορών κρατών μελών και των διάφορων ευρωπαϊκών χωρών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Μαρτίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας ε, με πολύ χαρά αλλά και συγκίνηση. Εγώ ανήκω σε μία γενιά ε, και ξέρετε ως ε, αντιπρόεδρος του ε, Κοινοβουλίου και ως σοσιαλιστής αγωνιστής ανήκω σε μια γενιά που έδωσε τη δική της μάχη, το δικό της αγώνα για την ελευθερία και για την αξιοπρέπεια. Και τέτοιοι αγώνε δίνονταν και σε πολλέ αφρικανικές χώρες και στη δική σας χώρα. Και θα αναφέρω τρεις Πορτογάλους αδελφού με τους οποίους ε, εγώ συνύπαρξα και στη στιγμή το Μάριο Σορέ, τον κύριο Αλμέντα Σάντο, τον Αντώνιο Αλμέντα Σάντο και φυσικά το Μανουέλα Αλέγρε με όλους αυτούς ε, είχαμε ε, πάρα πολύ στενές ε, σχέσεις και μπορώ να σας πω με πολύ μεγάλη χαρά ότι αυτά που κάνατε εσείς ως έργο της κυβέρνησης μας οδηγεί στο να σκεφτούμε ότι είχαμε δίκιο στην αλληλεγγύη που δείχναμε τότε. Σε άλλες περιπτώσεις υπήρξαν ε, κάποιες ανησυχίες και κάποια σύγχυση, απογοήτευση αν θέλετε, αλλά όχι στην περίπτωση του δικού σας έργου μέχρι σήμερα. γιατί ακριβώς ε, ακολουθεί το έργο σας ε, αυτά που είχαμε επιθυμήσει κι εμείς. Και στη συνέχεια θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω ότι εμείς ε, θα υποστηρίξουμε τις δικές σας προσπάθειες. Αναφερθήκατε και στο ότι κάποιες χώρες ε, μπορεί να ποινικοποιηθούν ως προς τη συνεργασία επειδή τα έχουν καταφέρει καλύτερα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί πάρα πολύ και αφορά και κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να θέσουμε εδώ, γιατί δεν θα είναι δίκαιο οι χώρες που έχουν καταβάλει τις μεγαλύτερε προσπάθειες και είχαν τις ε, μεγαλύτερες επιτυχίες ε, τελικά ε, να ποινικοποιηθούν ε, στα πλαίσια της συνεργασίας ε, και της υποστήριξης που θα έπρεπε να δοθεί από εδώ. Θα ήθελα να σας πω όχι ως κριτική, αλλά ως παρένεση. Και βασιζόμενος σε όσο είπε η Πορτογαλίδα συνάδελφος, εγώ θα ήθελα το πράσινο κροτήρι να διαδραματίσει έναν πιο ενεργό ρόλο στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής συνέλευσης των χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι εσείς μπορείτε να διαδραματίσετε ένα σημαντικό ρόλο και αυτή τη στιγμή δεν τον διαδραματίζετε με την ένταση που θα ήθελα εγώ. Αυτό το λέω γιατί ξέρουμε ε, το, ότι το πράσινο κροτήρι στο Συμβούλιο Βορρά Νότου, όπου είναι μέλος, έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και θέλω να παραθέσω και τον κύριο Μπαρόσο, άλλοι τον έχουν ε, γνωρίσει και ως Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, όμως εγώ τον γνώρισα ε, ως πρόεδρο αυτής της Επιτροπής συνεργασίας σε αυτή την Επιτροπή, σε αυτό το Συμβούλιο, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και εγώ νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσετε το ρόλο σας εκεί, σε αυτό το κοινοβουλευτικό όργανο. Και θα ήθελα να σας πω ότι όταν ακούσαμε τη Σεσάρια Εύωρα ε, να τραγουδάει, νοηρευόμασταν τη δημοκρατία και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας υποδεχόμαστε εδώ σαν αδελφό σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πισέπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά ε, σας υποδεχόμαστε σήμερα. Ε, σημείωσα όλες τις προόδους ε, στις οποίες αναφερθήκατε για τη χώρα σας είναι αρχιπέλαγος η χώρα σας. Ε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι θα πει αρχιπέλαγος, γιατί και εγώ έρχομαι από ένα αρχιπέλαγος από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, στους οποίους ε, έχετε ακόμη πολλή δουλειά ακόμη να ολοκληρώσετε, να ολοκληρώσετε και μιλάω για την ε, επισητιστική σας ανεξαρτησία. Ποιος, ποιους τρόπους έχετε προβλέψει, ποια μέσα προκειμένου να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση και κατά πόσο αυτό αποτελεί στόχο σας. Η ανάπτυξη της χώρας σας συνοδεύτηκε σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική ανάπτυξη. Ο τουρισμός βασίζεται ιδιαίτερα βέβαια σε οικονομικές συγκυρίες, οι οποίες μερικές φορές είναι ευμετάβλητες και θα ήθελα να μάθω, εκτός από την οικονομία του τουρισμού και τις γνώσεις που προσπαθείτε να αναδείξετε στη χώρα σας, Ποιες ε, είναι οι μεγάλες οδοί, ε, οι αναπτυξιακές που πιστεύετε ότι θα επιτρέψουν στη χώρα σας όχι μόνο να συνεχίσουν το δρόμο της πρόοδου, αλλά να ε, ολοκληρώσετε κάποτε τον αγώνα σας που τον έχετε ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, πράγμα για το οποίο σας συγχαίρω. Πρόεδρος, Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην, εξωτερική, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης. Ε, κύριε Ντόελ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, γιατί δυστυχώς έχει ενηλυμένες υποχρεώσεις ο πρόεδρος του Πράσινου Κροτηρίου και στις 5 η ώρα το αργότερο πρέπει να αποχωρήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ εκπροσωπώ την ε, κυρία Κάθριν Άστον. Θέλω να πω πόσο ικανοποιημένοι είμαστε που βρίσκεστε στις Βρυξέλλες και σας καλωρίζουμε εδώ και διαπιστώνουμε τις στενές σχέσεις μεταξύ της χώρας σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, είμαστε πολύ ευχαριστημένη με τις μεγάλες πρόοδους που έχει επιτύχει η χώρα σας. Όπως ε, βλέπετε κύριε Πρόεδρε υπάρχει ένας έξοχος συμβολισμός από τις δύο σημαίες που υπάρχουν πίσω σας οι οποίες μοιάζουν τόσο πολύ της χώρας σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2007 έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Καταρχάς έχουν τη μορφή της Σύμβασης για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και των επανεισδοχών που είναι αξιοσημείωτο γεγονός και όχι τόσο σύνηθες και επίσης έχουμε τη συμφωνία στον τομέα της ασφάλειας και σταθερότητος. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε μια πρώτη συνεδρία εργασία των δύο αυτών ομάδων στις Βρυξέλλες. Πέραν αυτού διαβλέπουμε μια εμβάθυνση των σχέσεών μας όσον αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα, τη μετανάστευση, τη τεχνογνωσία και την περιφερειακή ολοκλήρωση. Έχουμε, ε, ε, έχουμε ε, τακτικές διμερείς συναντήσεις. Συναντήσαμε τον Υπουργό Οικονομικών τον Οκτώβριο, τον Πρωθυπουργό τον, τον Νοέμβριο και την ετήσια διυπουργική διάσκεψη προς το τέλος του επόμενου έτους. Όλες αυτές οι διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις μας δίνουν την ευκαιρία να διαπιστώσουμε τη συνεργασία μας, τα διάφορα πλαίσια συνεργασίας. Επίσης έχουμε ε, συνεργασία, ενδελεχή συνεργασία στο θέμα της ασφάλειας στη Δυτική Αφρική και στην καταπολέμηση ε, πολλών δεινών που απειλούν την περιοχή, ναρκωτικά, βίες συγκρούσεις κλπ. Παρακαλώ ολοκληρώστε, ζήτησε η Πρόεδρος. Ε, θέλουμε λοιπόν μαζί να συνεργαστούμε για να αυξήσουμε το δυναμικό, να αναπτύξουμε το ανθρώπινο δυναμικό και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη των υποδομών. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Πρόεδρο του Πράσινου Ακροτηρίου για να απαντήσει στις παρατηρήσεις και στα σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω λίγα λεπτά στη διάθεσή μου και θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο τη δυνατόν ε, με μεγαλύτερη ακρίβεια στα σχόλια και στις ερωτήσεις που έγιναν. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτίνες ε, για τα πολύ φιλικά λόγια που μου απίφθηνε. Έφερε στο η μνήμη μου τη Σεζαρία Εύωρα και συντρόφους ε, αγώνων για την ανεξαρτησία, για την ελευθερία. Αναφέρεται και ονόματα που γνωρίζω σχετικά καλά. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω το εξή. Συμφωνώ μαζί σας για το ότι το πράσινο κροτήρι θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν πιο ενεργό ρόλο σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν πιο ενεργό ρόλο στην Αφρικανική Ένωση, στη CDO. Αλλά επίσης συμφωνώ και για την ε, συνέλευση στην οποία αναφερθήκατε. Θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα πιο σημαντικό ρόλο στη συνέλευση χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. θα τα θυμάμαι αυτά που υπόθηκαν ε, για να, για να μεταβιβάσω αυτό το μήνυμα. Εδώ βρίσκεται και ο κύριος ε, Σάντος, ε, ο οποίος άκουσε αυτές τις κριτικές που ακούστηκαν και να είστε βέβαιοι ότι θα βάλουμε τη δυνατά μας για να ενισχύσουμε το ρόλο μας εκεί. Όμως πολλές φορές μας λείπουν ε, τα μέσα. Πολλές φορές θέλουμε να συμμετάσχουμε πιο ενεργά, αλλά δεν έχουμε τα μέσα για μια πιο ενεργή συμμετοχή. Ακόμη και σε διμερείς ε, σχέσεις, ε, μια χώρα όπως το πράσινο ακροτήριο, όταν θα επιλέξει που θα ανοίξει μια πρεσβεία, πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά. Γιατί δεν έχουμε τα μέσα να ανοίξουμε παντού πρεσβείες. Μας λείπουν πόροι. Όμως, εγώ καταγράφω την ανησυχία σας και την πρότασή σας. Θα τη σκεφτώ. για τον κύριο βουλευτή που πήρε πρώτος το λόγο, δεν θυμάμαι το όνομά του. Έθεσε κάποια πολύ ενδιαφέροντα προβλήματα. Ποια θα είναι η φύση αυτής της προνομιακής εταιρική σχέσης στο μέλλον. Εμείς, όταν μπήκαμε σε αυτή την προνομιακή εταιρική σχέση το 2007, ίσως να μην γνωρίζαμε με ακρίβεια σε τι θα μπορούσε να μεταφραστεί. Είναι ουσιαστικά και ένα είδο δική μας μαθητείας. δηλαδή στο πώς να σχετιζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια αυτή τη ειδική σχέσης, τη προνομιακή σχέση. Μέχρι τώρα είχαμε την ενεργοποίηση των πόρων για την αναπτυξιακή συνεργασία. Όμως εμείς σήμερα στη συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο ε, της Επιτροπής, τον κ. Μπαρόσο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είδαμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε και άλλα μέσα και τρόπους συνεργασίας. Συζητήσαμε το θέμα της ασφάλειας και της σταθερότητας. Εμείς θέλουμε να είμαστε μια χώρα χρήσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να είμαστε ένας εταίρος αξιόπιστος και σίγουρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένως, όταν εμείς δείχνουμε διαθέσιμοι να συνεργαστούμε σε θέματα ασφάλειας, στους ε, θαλάσσιους διαδρόμους του Ατλαντικού για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και συναφών φαινομένων, εμείς Θέλουμε μεν να είμαστε χρήσιμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε να υπερασπίσουμε και τα δικά μας συμφέροντα ως κυρίαρχη χώρα και ως δημοκρατία, ως κράτος δικαίου, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Όμως, επίσης, σκεφτόμαστε και κάποιους άλλους τομπείς Ίσως ε, θα πρέπει να σκεφτούμε και πώ θα στηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα στο πράσινο ακροτήρι. Γιατί μια οικονομία όπω η δική μα, που είναι μια οικονομία υπηρεσιών, και ξέρετε ότι μια τέτοια οικονομία για να είναι βιώσιμη πρέπει να δημιουργήσει συνθήκε για να αυτοχρηματοδοτήσει την αναπτυξιακή της διαδικασία. Έτσι λοιπόν, για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί ο ιδιωτικό τομέα. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης μπορεί να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Ο κύριος Μπαρόσο είπε σήμερα και εμείς συμφωνούμε ότι ίσως να υπάρχουν περιποθέσεις για να ενισχύσουμε να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε μία σύνδεση Ευρωπαίων επιχειρηματιών με επιχειρηματίες από το πράσινο κροτήρι. Αλλά έχουμε κατά νου και τομεί όπως οι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Οι τομεί όπως ε, αυτή στους οποίους αναφέρθηκε η κυρία Καρβάλιο. Καινοτομία, η επιστήμη, νέες τεχνολογίες, η ανωτατή εκπαίδευση και η έρευνα. Και εγώ πριν να γίνω πρόεδρος, ξέρετε, ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Και ουσιαστικά ήμουν διευθυντής, μου άνοιγε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο Πράσινο Κροτήρι. Όμως εμείς στο Πράσινο Κροτήρι ονειρευόμαστε να γίνουμε μία αναπτυγμένη χώρα. Θέλουμε να πάμε πιο πέρα και μια χώρα δεν μπορεί να πετύχει την ανάπτυξη αν δεν έχει υψηλή εξειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να έχουμε ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, αλλά το πόσο μάλλον στην ανώτατη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μπορεί επίσης να είναι ένας τομέας που θα ενισχυθεί από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των ερευνητών, μεταξύ των ε, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να ενισχύσουμε ένα δίκτυο που θα χρησιμεύσει και στο πράσινο ακροτήρι, αλλά και σε γειτονικές χώρες. Εγώ, παραδείγματος χάρη, Έχω κατά νου την περιφέρεια της Δυτικής Αφρικής ε, ή ε, την κοινότητα των Πορτογαλόφωνων χωρών. Υπήρξε και κάποιος άλλος ε, ομιλητής που αναφέρθηκε στο θέμα της επιτιστικής ανεξαρτησίας, στον τουρισμό. Ναι, βέβαια, ο τουρισμός είναι ένας ζωτικός τομέας για μας. Στο πράσινο κροτήρι. Υπάρχει μια συνένεση από όλα τα πολιτικά κόμματα και από τους ειδικού όλων των τομών ότι ο τουρισμός στο πράσινο ακροτήρι πάντοτε θα είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας όμως προφανώς υπόκειται σε διακυμάνσεις και επηρεάζεται από εξωτερικές εξέλιξεις. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε και συμπληρωματικές οδούς ανάπτυξης. Παραδείγματος χάρη ο τομέας ε, της ανάπτυξης της γεωργίας ε, και της κτηνοτροφίας. Ο γεωπισητιστικός τομέας, όπως λέγεται, πρέπει να βελτιωθεί για να βελτιώσουμε και τα επίπεδα της επιστημικής μας ανεξαρτησίας, αλλά και σε συνεργασία με τον τομέα του τουρισμού. Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε μια χώρα που αποτελεί μια πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών προς το εξωτερικό στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, στον τομέα των ε, θαλάσσιων μεταφορών, των νέων τεχνολογιών, πληροφοριών και γενοτομίας. Και γι' αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε, βασιζόμαστε στην συνεργασία με οργανισμούς όπως η ΦΑΟ, αλλά όπως ε, και η κοινότητα των πορτογαλόφων χωρών ε, και σε εκείνο τον οργανισμό η πιστιστική ανεξαρτησία έχει λάβει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα σε μια σύνοδο κορφής ε, που έλαβε χώρα πρόσφατα. Εγώ θα κλείσω λέγοντας το εξή. επαναλαμβάνοντας. Εμείς ε, σκεφτόμαστε στο πράσινο κροτήρι ότι πρέπει να έχουμε τη διάβια αλλά και τη δημιουργικότητα και τη φαντασία για να επαναφεύρουμε κάθε στιγμή αυτήν την προνομιακή εταιρική σχέση χωρίς ε, όρια. Μάλλον το όριό μας ε, είναι να γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια αυτό δεν είναι δυνατόν, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ένθερμη υποδοχή σας εδώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εξ ονόματος των δύο επιτροπών μας, ε, Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελα να σας διαβάσω τις πιο θερμές ευχαριστίες για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα προχωρήσουμε σε τρεις σύντομες ε, ψηφοφορίες της Επιτροπής Ανάπτυξης. Και μετά από τις ψηφοφορίες αυτές και πάλι θα περάσουμε στο από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σημείο σχετικά με την κατάρτιση της κατάστασης με τους τρεις υποψηφίους για το βραβείο Ζαχάροφ. παρακαλώ πολύ ε, έχετε διαθέσιμες τις ε, κάρτες ψηφοφορίας να κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Άρχεται η ψηφοφορία. Voilà, tout le monde pas Δεν ψήφισαν ακόμη όλοι. Πέντε ψήφοι, λοιπόν. Έξι. Παρακαλώ, βγάλτε τις κάρτες σας. Ωραία. Ψηφίσατε όλοι. Ο κύριος Μπρόκ δεν ψήφισε. Σχόλιο από την αίθουσα. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. για τη δική μας συνεισφορά σε σχέση με την επιστημιστική ασφάλεια και τα κλιματικά εν ώψη της διάσκεψης στη Φαρσοφία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Όχι, λέει η Πρόεδρος, συμβιβαστική τροπολογία, απλώς, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Ωραία. Ελέγχουμε τροπολογία 6. Το δεύτερο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Είναι υπεράριθμο το ΕΛΚ. Κύριε Μπρόκ, μήπως δεν πρέπει να ψηφίσετε.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 εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατά τμήματα ψηφοφορία, τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Α, καταπίπτει λέει η πρόεδρο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τροπολογία 13, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. να ψηφίσουμε όλες μαζί τις τροπολογίες από 15 μέχρι 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Θα ήθελα ένα διαδικαστικό, λέει ο κύριος Μίτσελ με ενημερώνουν ότι μόνο 10 ψήφους είχε το ΕΛΚ, ε, άρα ο κύριος Μπροκ μπορεί να ψηφίσει. Εδώ, αυτό μου λένε ε, το προσωπικό της ομάδας. Ωραία. Ας το κάνουμε τότε ηλεκτρονικά. Θα αφήσουμε όλους τους συναδέλφους του ΕΛΚ να ψηφίσουν ηλεκτρονικά για να δούμε τι γίνεται. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρα της Άρα μπορείτε να ψηφίσετε κύριε Μπρόκ. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 19, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20, πάλι κατά τμήματα ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στο δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Λείπουν τέσσερις ψήφοι. Πέρα τη ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Κυρία Πρόεδρε, πάλι ο κύριος Μίτσελ, διαδικαστικό, συγγνώμη που καθυστερώ τη συνεδρία σας, αλλά το γεγονός ότι δεν ε, μπόρεσε να ε, ψηφίσει ο κύριος Μπρόκ, ε, μήπως επηρεάζει τις υπόλοιπες ψηφοφορίες, όχι ήταν πολύ μεγάλη διαφορά, λέει η Πρόεδρος. Ωραία. Ψηφίζουμε τώρα την τροποποιημένη γνωμοδότηση, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και θα ψηφίσουμε τώρα και ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Ωραία. 27 υπέρ, 3 ε, κατά και καμία αποχή. Ψηφίζουμε τώρα την γνωμοδότηση κορτέ Λάστρα. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, α, καταπίπτει. Πάμε τώρα στο τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροποποιηθήσα γνωμοδότηση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε και ηλεκτρονικός όμως, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 28 υπέρ, 25 κατά, ε, συγγνώμη, 3 ε, κατά. Ε, και πάμε τώρα στην τελευταία ψηφοφορία για την έκθεση Bill Newton Dunn. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος, ε, ήταν δύο τμήματα. Οπότε θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Και δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω σε ποια χρονική στιγμή σηκώσατε το χέρι στο υπέρ ή στο κατά. Ξαναρχίζω λοιπόν. Υπέρ. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30, 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 Α, έλεγχος. Έλεγχος θέλετε τη 40. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την τροπολογία 40. Λοιπόν, δύο υπεράριθμοι στο ΕΛΚ. Ένας για τους σοσιαλδημοκράτες και δύο για τους φιλελεύθερους. Λοιπόν, ψηφίζουν τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης. Εντάξει. Λοιπόν, ξαναρχίζουμε. Λοιπόν, στους αντιδημοκράτες είναι υπεράριθμοι κατά έναν. Ένας παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Κύριε Μπρόκ, μάλλον πρέπει να μην ψηφίσετε, γιατί πάλι έχουμε έναν παραπάνω στο ΕΛΚ. Κύριε Μπέρμαν, μήπως μπορείτε εσείς να μην ψηφίσετε. Ποιος δεν θα ψηφίσει από τους σοσιαλδημοκράτες. Κύριε Μπέρμαν, μπορείτε να βάλετε τάξη στην ομάδα σας. Ένας παραπάνω είναι που ψηφίζει. Το ξαναλέω, είναι ένας παραπάνω στους σοσιαλδημοκράτες. Λοιπόν, αποφασίσατε. Α, εντάξει τώρα. Λοιπόν, άρα, ελέγξαμε τροπολογία 40. Πέρας. Ε, δεν είναι δυνατόν αυτό το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 42 συγγνώμη απορρίπτεται 42 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ. Α, πρέπει να ψηφίσουμε και την 60, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος της 65. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60... 7. Όχι, 68 διερθώνει η πρόεδρος, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 69, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος της 74 έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 77. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Όχι, καταπίπτει. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Καταρχάς με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα και ηλεκτρονικός. Έναρξη ψηφοφορίας. Ένας από τους σοσιαλιστές να μην ψηφίσει. Είστε υπεράριθμοι κατά έναν. Α, εντάξει τώρα. Ωραία. Πέρασα. Της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος ε, κατά και 5 αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Υπάρχουν άλλα ερωτήματα για, για τα μέλη της Επιτροπής μας. 3 Οκτωβρίου, 9 ε, και 35 η επόμενή μας συνεδρίαση και στις 14 ε, το απόγευμα. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην ε, από κοινού μας συνεδρίαση με την Επιτροπή